Уважаеми колеги, за Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προνόμιο για μένα, αλλά και με μεγάλη χαρά συμπροεδρεύω σήμερα εδώ στην συνεδρίασή μας αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη στη σταθερότητα, τον οικονομικό συντονισμό και την διακυβέρνηση. Βάλτε τα ακουστικά σας, ε, αν θέλετε να καταλάβετε τα βουλγαρικά. Τα είπα μέχρι τώρα, βουλγαρικά, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καλωσορίζω όλους σας εδώ και την κυρία Τάισεν βέβαια που δέχτηκε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή. Το πρώτο τμήμα έχει να κάνει με τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018. Θα συζητήσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες λοιπόν του εξαμήνου αυτού, έτσι όπως αναφέρονται στην έκθεση για την σταθερότητα και την ανάπτυξη που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα έχουμε και τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας των Επιτροπών Οικονομικών και την Κοινωνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συγητές τους θα μας ενημερώσουν για το πώς προχωρούν οι εκθέσεις αυτές μέχρι σήμερα. Θέλω να ζητήσω επίσης συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Γκουαλτιέρη, ο οποίος δυστυχώς ε, πήγε σε μια συνεδρίαση η οποία κράτησε περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι εδώ στην αρχή, αλλά θα έρθει σε λίγο για να συμπροεδεύσει μαζί μου. Οι διάφορες αντιπροσωπείες θα θέλαμε να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους και να μας πούνε πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαστούμε για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Θέλω επίσης να σας πω δύο λόγια για το πόσο θα οργανωθεί η συνεδρίασή μας αυτή. Λοιπόν, υπογραμμίζω ότι για να πάρετε το λόγο στη συνεδρίαση αυτή. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όσοι ήθιστε θα φροντίσουμε όσο γίνεται περισσότεροι από αυτούς που θέλουν να πάρουν το λόγο, όντως να πάρουν το λόγο για να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ακόμα και αν ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένος. Και επειδή είναι πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετοχόντων, σας παρακαλώ δείξτε κατανόηση και πολύ πιθανόν δεν θα είναι δυνατόν όλοι σας να πάρετε το λόγο. Γι' αυτό και σας ζητώ επίσης να περιοριστείτε σε ένα με δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σας, το πολύ. Θα υπάρχει το ρολόι, θα το βλέπετε στην οθόνη. Και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε το χρόνο για να τηρήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα, γιατί όπω ξέρετε, μετά από αυτή τη συνεδρία ακολουθούν και άλλε. Στα να σα θα βρείτε τι κάρτε τι οποίε πρέπει να συμπληρώσετε για να ζητήσετε το λόγο. Αν θέλετε το λόγο, τότε συμπληρώστε τις κάρτες αυτές και δώστε στους κλητήρες, οι οποίοι κυκλοφορούν στο ημικύκλιο. Αυτό ισχύει τόσο για τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, όσο και για τους ευρωβουλευτές. Γενικά μιλώντας θα προσπαθήσουμε το χρόνο ομιλίας να τον κατανοήμω ως εξής. Τρεις εθνικοί βουλευτές, ένας ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Αν χρειαστεί να αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, θα το κάνουμε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η Βουλγαρική Προεδρία δεν είναι μεγάλη σημασία στην κοινοβουλευτική διάσταση τα εθνικά κοινοβούλια στις χώρες τους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την λογοδοσία των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των πολιτών της. Έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά, επίσης τα δημοσιονομικά των χωρών μελών. Υπάρχει μια βελτίωση και πιστεύω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια, όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να φροντίζουν για πολιτικές που θα στηρίξουν μεταρρυθμίσεις για να προωθηθεί το θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο, να δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης ποιότητα και να μειωθούν οι ανισότητες. Και πάλι λοιπόν, εκ μέρους της Βουλγαρική Προεδρίας, σας καλωσορίζω εδώ και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Τάισεν. που είναι Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, επαγγελματικών ε, προσόντων και κινητικότητα στον χώρο τη εργασία. Παρακαλώ κύριε Τάση να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα αλλά και μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στι μεταρρυθμίσει και στη βελτίωση των οικονομιών μα αλλά και των κοινωνιών μα. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Και είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα γιατί μετά από αρκετά χρόνια κρίσης είναι ωραίο να μπορεί κανείς να φέρει ωραία νέα. Η ανάπτυξη έχει επανέλθει σε όλες τις χώρες μέλη. Υπάρχει ανάκαμψη των επενδύσεων επίσης και υπάρχει και περισσότερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα από ό,τι παλιότερα. Βέβαια, δεν έχουμε ανακάμψει πλήρως από την οικονομική κρίση. Ακόμα έχουμε υψηλά επίπεδα ε, χρεών, τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. Πάνω από δεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άνεργοι και βλέπουμε τέτοια φαινόμενα σε όλες τις χώρες μέλη. Συνεπώς, ο πρώτος στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι η ανανέωση αυτή στην ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ότι δηλαδή θα πετύχουμε σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι οικονομίες μας, οι κοινωνίες μας είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που υπάρχουν και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Jean-Claude Juncker, είπε ότι τη σκεπή τη φτιάχνει κανείς όταν κάνει καλό καιρό και όχι με κακοκαιρία. Συνεπώς, τώρα προετοιμάζουμε τις εκθέσεις αναχώρα για να είναι έτοιμες στις 7 Μαρτίου. Πρόκειται για την ανάλυση των κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική των διαφόρων χωρών που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια το Μάιο. Οι εκθέσεις αναλύουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τις τάσεις που κρατούν στις χώρες μέλη και γίνεται και επίσης αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών αναχώρασης στάσεων του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν θα ήθελα σήμερα μαζί σας να μοιραστώ το μήνυμα που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, Ας ε, χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρα στις μεταρρυθμίσεις μας. Πηγαίνουμε όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Από τότε που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το 2011 δηλαδή, οι χώρες μέλη έχουν επιδείξει πρόοδο όσον αφορά τα δύο τρίτα των συστάσεων τουλάχιστον. Και στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος ή υλοποιήθηκαν πλήρως οι συστάσεις. Δεύτερον, η σύγκληση η οποία υποχώρησε κατά τη διάρκεια της κρίσης, τώρα επανέρχεται. Υπάρχουν θετικές προοπτικές λοιπόν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη. Όμως δεν υπάρχει περιθώριο για να αναπαθούμε. Οι ανάγκες παραμένουν. Οι ανισότητες μάλιστα έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες μέλη. Αν λοιπόν δεν αλλάξει η κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόκληση θα είναι τεράστια και θα κινδυνεύει η ίδια η συνοχή. Έπειτα, η συνολική έκθεση των τραπεζών έχει μειωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες. Υπάρχει ανάκαψη σε όλες τις χώρες μέλη, όμως σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να υπάρχει πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος, από το οποίο κινδυνεύουν οι συλλογισμοί των τραπεζών και επενδύσεις βέβαια. Και σε μερικές χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν ε, μεγάλα και πολλά δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα. Οι συνθήκε στην αγορά επίσης βελτιώνονται, η δουλειά όμως δεν έχει τελειώσει. Η ανεργία, ο κίνδυνος της φτώχειας παραμένουν. Τα νούμερα είναι ιδιαίτερα υψηλά σε πολλές χώρες μέλη. Και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος ανεργίας μεγάλος και η διαφορά των ορών που εργάζονται οι εργαζόμενοι ε, διαφέρει όλο και περισσότερο από χώρα σε χώρα. Όμως το πιο σημαντικό μήνυμα του εξαμήνου είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος πάνε χέρι-χέρι. Οι επενδύσεις στον κόσμο είναι αυτό που οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, ισότιμες κοινωνίες βοηθούν την ανάπτυξη. Μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν να έχετε το αναχωριστό άλλον. άλλο. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά είναι τρεις διαστάσεις οι οποίες πρέπει να προχωρούν παράλληλα. Και αυτό είναι και εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έγινε πιο κοινωνικό. Ο φετινός κύκλος πάντως αποτελεί ορόσημο. Πριν από μερικούς μήνες ε, μιλήσαμε για τον κοινωνικό πυλώνα. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού είπανε ότι ο πυλώνας αυτός αποτελεί μια δέσμευσή μας για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη και ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Και ο πυλώνας αυτός ε, περιλαμβάνει διάφορα κοινωνικά δικαιώματα και δείχνει πού πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο όμω η επιτυχία του πυλώνα αυτού εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο θα υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. Αφού λοιπόν καταλήξαμε στην διακήρυξη του πυλώνα αυτού, προχωρούμε στις αρχές του πυλώνα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και για την υλοποίησή τους προχωρήσαμε σε ένα κοινωνικό βαθμολόγιο με 40 δείκτες προκειμένου να είμαστε σε θέση να κρίνουμε πώς προχωράμε σε αυτό το πυλώνα. Το βαθμολόγιο αυτό λοιπόν, τα κριτήρια αυτά θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις εκθέσεις αναχώρα και στις συστάσεις αναχώρα στη συνέχεια. Κοιτώντας την ανάλυση μας μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερις αρχές οι οποίες επανέρχονται στις συστάσεις μας. Πρώτον, δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη βελτίωση του ελλείμματος. Έχει σημασία και η ποιότητα των ε, δημοσίων δημοσιονομικών, τα φορολογικά συστήματα που πρέπει να είναι δίκαια, υπέρ της ανάπτυξης, να ενθαρρύνουν ε, την απασχόληση και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δεύτερον, η επένδυση στον άνθρωπο είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μόνο μορφωμένοι εργαζόμενοι με προσόντα μπορούν να βοηθήσουν στις αλλαγές που χρειαζόμαστε στην αγορά εργασίας και χρειάζεται και ασφάλεια για όλους τους εργαζόμενους γιατί μόνο τότε μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη μετάβαση στο νέο κόσμο της εργασίας. Τρίτον, χρειάζονται γενικότερα περισσότερες επενδύσεις γιατί οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις είναι κάτι πιο κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ΑΕΠ μας. Και έπειτα η ανάπτυξη οδηγεί στη μείωση των ανισοτήτων και διασφαλίζει υψηλά επίπεδα διαβίωσης. Χρειάζονται σωστά συστήματα και σωστοί μηχανισμοί. Είναι κάτι πολύ βασικό προκειμένου να διασφαλίσουμε ε, αυτήν την ε, διαφοροποίηση στους μισθούς. Όλα εξαρτώνται βέβαια από την κατάσταση στην κάθε χώρα και πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας και τις αλλαγές στην παραγωγικότητα. Όλα αυτά δεν είναι λίγα για τις χώρες που πρέπει να τελοποιήσουν, ούτε είναι εύκολο να καθοριστούν σωστά και με αξιοπρέπεια οι κανόνες. Θέλουμε αποτελέσματα με το λιγότερο κόστος. Θέλουμε να καταναμηθεί το βάρος ισότιμα. Θέλουμε να ακούγονται όλες οι φωνές και να υπάρξει ενστερνισμός των αποφάσεων και επίσης θέλουμε ε, μακροπρόθεσμα να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο ωφέλη. Ε, αγαπητοί συμπρόεδροι, κυρίες και κύριοι, οι εκθέσεις αναχώρα αποτελούν μόνο την αφετηρία της δεύτερης αυτής φάσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018. Όπως έγινε και πέρυσι, θα έχουμε άφθονο χρόνο για να συζητήσουμε με τις εθνικές κυβερνήσεις και με τις κοινωνίες συνολικά πριν γίνει η δημοσίευσή τους κάτι το οποίο μας βοηθάει να είμαστε πιο ακριβείς στην ανάλυση μας, αλλά επίσης βοηθάει τη διεξαγωγή διαλόγου και αμοιβαία κατανόηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και χώρες μέλη αποτελούν πολύ σημαντικό εταίρωμα στο διάλογο αυτό. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ε, πολλοί επίτροποι και εγώ προσωπικά θα ταξιδέψουμε και ταξιδεύουμε στις διάφορες χώρες μέλη για να συζητάμε με τους ομολόγους μας στις χώρες μέλη για όλα αυτά, όπως επίσης και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους. Κυρίε και κύριοι, πρόκειται για ένα κοινό εγχείρημα, μια κοινή αποστολή. Οι εκθέσεις αναχώρα λοιπόν ας αποτελέσουν την αφετηρία και εγώ ε, πραγματικά ε, βιάζομαι να ξεκινήσω το έργο μου μαζί σας για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε κυρία Τάισεν. Ανεκτήμητα τα σχόλιά σας. Ε, είμαι βέβαιη ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται για κοινή αποστολή. Δεύτερος ομιλωτής, ο κύριος Κρίστοφ Χέτβαν, ε, εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2018 από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. κύριε Χέτμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας όσον αφορά την ετήσια στρατηγική ανάπτυξης. Καταρχάς όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, ε, κύρια Επίτροπο και το Σώμα των Επιτερόπων που κατάρτισαν την ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη που αποτελεί και την πηξίδα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είμαστε βεβαίως πάρα πολύ χαρούμενοι που η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει. Υπάρχει αύξηση των επενδύσεων και μείωση της ανεργίας. Το ΑΕΠ είναι υψηλότερο από ό,τι περιμέναμε και εάν το εξετάσουμε από το πρίσμα των μακροοικονομικών, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Βεβαίως υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Παρά όλα τα θετικά στοιχεία, ε, συνειδητοποιούμε ότι ακόμα εκρεμούν πολλά. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι Ακόμα είναι πάρα πολύ υψηλή η ανεργία των νέων. Είναι πάνω από το 16% αυτή τη στιγμή. Πάνω από 16 εκατομμύρια ε, νέοι άνθρωποι ηλικίας 15 έως 24 ετών ε, ούτε εργάζονται ούτε φοιτούν ε, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και φυσικά υπάρχουν και πολύ υψηλά ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού και αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο. Για να μπορέσει να είναι επιτυχή η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξωμενού χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Καταρχάς με ακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις και δεύτερον θα πρέπει κάθε χώρα να λάβει υπόψη τις συστάσεις αναχώρα και να τις εφαρμόσει σωστά. Και αυτό είναι και το αδύνατο σημείο μας. Δεν γίνεται πολύ σωστά η εφαρμογή. Εάν δούμε τι έγινε το 2016... πλήρης εφαρμογή υπήρξε μόνο ε, στο 2% των συστάσεων, εν μέρη η εφαρμογή είχαμε στο 40%, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 55% των συστάσεων δεν εφαρμόστηκαν σχεδόν καθόλου. Το ερώτημα λοιπόν για μας είναι γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μήπως συμβαίνει διότι όπως επισημαίνει, ε, επισημαίνουν κάποιοι υπάρχουν προβλήματα με τα εθνικά θεσμικά όργανα ή γιατί τα κράτη-μέλη προτιμούν να εφαρμόσουν τις δικές τους λύσεις, τις δικές τους στρατηγικές για να επιλύσουν το πρόβλημα. Εκεί όμως τίθεται το ερώτημα ε, του κατά πόσον αυτά είναι συμβατά με αυτά τα οποία συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν εξετάσει κανεί τα στοιχεία, δυστυχώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο και μπορεί βέβαια και οι συστάσει να είναι πάρα πολλέ ή πάρα πολύ φιλόδοξε για κάποιε χώρε. Πρόκειται για κάτι το οποίο εκκρεμεί και πρέπει να διαπιστώσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και φυσικά πρέπει να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος. Βεβαίως αυτό που προέχει είναι να είμαστε ρεαλιστές. Ε, όσες φορές και να το πω δεν είναι αρκετές. Ε, πρέπει να έχουμε φιλοδοξία στους στόχους μας, αλλά θα πρέπει να είναι και εφικτή η εφαρμογή τους. Ε, πέρσι τον Νοέμβριο, στη διάρκεια της Κοινωνικής Συνέδου στο Γκέτεμπεργκ, τα τρία θεσμικά όργανα ενέκριναν τον ε, πυλώνα των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το έγγραφο αυτό απαριθμεί όλες τις αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία της αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Πιστεύω ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να αποτελούν σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής σύγκλησης στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και φυσικά θα πρέπει να θυμόμαστε και τις διαθεωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες στόχο έχουν να βελτιώσουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, θα πρέπει να υπάρχει ε, περιθώριο για υψηλότερους μισθούς και βεβαίως θα πρέπει να βελτιώσουμε και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό λοιπόν και ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Γεγονό το οποίο με οδηγεί σε ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο πλήττει πάρα πολλού πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και πέρσι το Μάρτιο. Κατά τα φαινόμενα, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, οι ανισότητες ε, στα εισοδήματα αυξήθηκαν ε, στα δύο τρίτα των κρατών μελών. Αυτό βεβαίως ε, συμβαδίζει και με υψηλά ποσοστά ανεργίας ή ε, πολύ επισφαλείς ε, συμβάσεις στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα είναι ότι τόσο όσον αφορά τους μισθούς αλλά και όσον αφορά τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών, και εδώ φυσικά δεν αναφέρομαι απλώς στα παλιά ή στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι καθολικό και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το χάσμα διευρύνεται και ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μειώνεται. Και εδώ έρχεται να προσθεθεί και ένα ακόμα πρόβλημα, ενδοπεριφερειακές διαφορές, οι οποίες εντείνονται όλο και περισσότερο. βλέπουμε το ένα τμήμα της περιφέρειας να γίνεται φτωχότερο και το άλλο τμήμα ταυτόχρονα να γίνεται πλουσιότερο. Υπάρχει βεβαίως η πολιτική συνοχή που είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και επομένως πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να υπάρχουν μέτρα στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά ε, δεν θα αποτελέσει και πανάκια για όλα μας τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε ε, μια πολιτική συνοχή πολύ πιο φιλική προς το χρήστη, με πολύ λιγότερη γραφειοκρατία και πολύ πιο κοντά ε, στον τελικό δικαιούχο. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και αυτό που χρειάζεται η αγορά εργασίας. Πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν στις ψηφιακές γνώσεις της κοινωνίας μας. Το 90% όλων των θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες στην αγορά εργασία ε, προϋποθέτουν και κάποιες ψηφιακές γνώσεις. Και πάρα πολλοί άνθρωποι στην αγορά εργασίας, περίπου το 43%, δεν φαίνεται να διαθέτει αρκετά προσόντα όσον αφορά τις ψηφιακές αυτές δεξιότητες. Ε, οι εργοδότες επισημαίνουν ε, συνεχώς ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να καλύψουν αυτά τα οποία αναζητούν. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και η κατάλληλη σχέση μεταξύ εργοδότη εργαζομένου. Είναι αρκετά υψηλή η ανεργία μεν, αλλά οι εργοδότες φαίνεται ότι δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους. Και φυσικά αυτό συμβαδίζει και με την ανταγωνιστικότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές σε αυτό το τομέα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη κατά τρόπον ώστε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να άρουμε όλα τα προσκόμματα για τη δραστηριοποίησή τους στην αγορά. Και εδώ φυσικά η πολιτική συνοχή θα μπορούσε να βοηθήσει και μάλιστα όχι μόνο αυτούς που θέλουν να επενδύσουν σε καινοτόμες δεξιότητες και σε καινοτόμες λύσεις, αλλά και εκείνους που απλώς επιθυμούν ε, να ε, μορφώσουν καλύτερα τους μαθητές μας. Επίσης, ε, ε, νέες δεξιότητε για νέε υπηρεσίε. Προφανώς και η καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντική και μία από τις πιο σημαντικές και τελευταίες πολιτικές προτεραιότητε που θα ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι η κοινωνία μας γυράσκει και οι άνθρωποι φεύγουν ε, από τις ε, μεθοριακές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου. Αν δούμε τον πληθυσμό της υπαίθρου, βλέπουμε ότι οι ανθρώπινοι πόροι κινούνται μόνο προς μία ε, κατεύθυνση. Οι περιφέρειες ε, ε, στις αστικές περιοχές ε, είναι όλο ένα και πιο ε, πολυπληθείς και οι άνθρωποι γίνονται όλο και φτωχότεροι. Επομένω θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες και πώς μπορούμε να προσφέρουμε και πιο ευέλικτες λύσεις για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε και τα συνταξιοδοτικά συστήματά μας, ε, να μην εξετάζουμε τόσο την ηλικία συνταξιοδότησης όσο τον αριθμό των ετών ε, που κάποιος συνεισφέρει στα ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ η ετήσια έκθεση ανάπτυξης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα και όλα αυτά τα επιχειρήματα από όλε τι πλευρέ. Εγώ όμω είμαι αισιόδοξο και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε όλα και ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα αποτελέσει ένα στεναρό μήνυμα και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χέτμαν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ομιλητές ότι χρειάζεται, είναι ανάγκη να μιλούν πέντε λεπτά το πολύ για να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χιου Μπαγιέ, που είναι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τον, τον οικονομικό συντονισμό. Έχετε πέντε λεπτά, κύριε Μπαγιέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Λοιπόν, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που έχουμε, που είναι ακόμα βέβαια διστακτικά, αλλά είναι θετικά στην Ευρωζώνη. Όμως οι μακροοικονομικοί δείκτες δεν οδηγούν στην κατάργηση των ανισοτήτων μέσα στην ίδια χώρα, δεδομένου ότι έχουμε εργαζόμενους ακόμα φτωχού και δεν υπάρχει σύγκληση μεταξύ των χωρών μελών. Σε αυτό βασιστήκαμε για να διαπραγματευτούμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το κείμενό μας, το οποίο πρέπει να ψηφιστεί τώρα την ε, Τετάρτη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βανκίντελάρ και τον κύριο Λουλίκ που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα, που είναι οι συνεισηγητέ μου, οι σκιώδει συνεισηγητέ ουσιαστικά. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει ένα κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο το οποίο να είναι σταθερό και όπως είπε και η Επίτροπος να οδηγήσει σε απασχόληση η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Όπως επίσης γνωρίζετε οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ε, το αδιέξοδο των ε, γρήγορων αλλαγών στον, στην αγορά εργασίας χωρίς να προλαβαίνουν να προσαρμοστούν. Γι' αυτό και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θέλαμε ένα κεφάλαιο που να αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά μας, στην έρευνα ε, και την ανάπτυξη στην Ευρώπη, στην ψηφιακή τεχνολογία, επιμένοντας στο να, δοθούν, ε, στο να δοθεί βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην νεολαία, μέσω πολιτικής ε, κατάρτισης, αλλά και διαβίου μάθησης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Επίσης, να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητα των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Όπως το είπε και η Επίτροπος, υπάρχει πλέον ο πίνακα με τα κριτήρια, το βαθμολόγιο κατά κάποιο τρόπο, οπότε μπορούμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε αφιερώσει και ένα κεφάλαιο τη έκθεσής μα στην αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία. Όπω γνωρίζετε, στι ιδιωτικέ ε, επενδύσει έχουμε επανέλθει σε ίσα στα επίπεδα του 2008 ενώ για τις δημόσιες επενδύσεις βρισκόμαστε ακόμα πολύ πιο κάτω. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει, να δει ποια είναι τα εμπόδια στα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Αυτά τα επενδυτικά προγράμματα συνήθως ε, βέβαια είναι συνδυασμό, συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Τι είναι αυτό που αποτελεί τροχοπέδι λοιπόν, γιατί δεν ξεκινούν τέτοιες επενδύσεις ξανά. Έπειτα υπάρχει και το θέμα της ε, φορολογικής αναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε από την αρχή της θητείας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και κυρίως η Οικονομική μας Επιτροπή. Ξέρουμε ποια είναι η φορολογική κατάσταση στις χώρες μέλη που επιτρέπει σε διάφορες πολυεθνικές να επιλέγουν ε, τη χώρα που τους συμφέρει περισσότερο. Αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός πρέπει να σταματήσει προς όφελος των πολιτών μας και των χωρών μας. Θέτουμε επίση και το θέμα της αύξηση των μισθών. Είναι μια πρόταση που έχει στηρίξει και ο Μάριο Τράγκη ώστε να υπάρξει περισσότερη αγοραστική δύναμη στους εργαζόμενους και στα νοικοκυριά. Πιστεύουμε ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν θετικά και αποτελεσματικά μέτρα και να μειωθούν επίσης και τα βάρη στις δημόσιες δαπάνες. Και κάτι άλλο είχε να κάνει με, τον, με τι κατευθύνσεις γραμμέ του προπολογισμού που πρέπει να επιτρέψει τη βιωσιμότητα των δημοσίων δαπανών και καλή διαχείριση αυτών. Όπω και ο συνάδελφο από την Επιτροπή Επασχόληση, και εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια στι συστάσει. Πρέπει να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με περισσότερη διάδραση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην οικονομική και κοινωνική πολιτική των χωρών μα. Ελπίζουμε το Σεβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν υπόψη του τι νέε αυτέ κατευθυντήριε γραμμέ που προτείνουμε και ελπίζουμε την Τετάρτη να πετύχουμε ικανοποιητική συμφωνία Προ όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπαγιέ. Πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Μιλόσεβιτς, τον επόμενο μιλητή. Θα ήθελα να, ευχα... ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους τη Βουλευτικής Αντιπροσωπείας, η οποία έχει ε, συνάντηση με τον κύριο Ταγιάννη και την ε, πρόεδρο του, της ε, Βουλγαρικής Βουλής. Χωρίς περαιτέρω χρόνο τριβή, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιβάν Μιλόσεβιτς, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κροατικού Κοινοβουλίου. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο, κύριε Μιλόσεβιτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Βουλγαρική Προεδρία για την πρόσκληση που απίφθηνε σε εμάς. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, όπως είναι η ανάκαψη, η απασχόληση ε, και η ευημερία. Θα ξεκινήσω με κάποια γενικά θέματα, συνέχεια θα αναφερθώ στη σύγκληση και μετά θα σας δώσω την κροατική οπτική. Προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, εγώ πάντοτε είμαι υπέρ της κατάργησης των δαπανών και της γραφειοκρατία. Όμως, ε, ο προϋπολογισμός σε σχέση με, με το ΑΕΠ της Ευρώπης δείχνει ότι αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες είναι οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε. Ένα άλλο ζήτημα. Η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών φορολογικών συστημάτων θα επηρεάσουν την, το παγκόσμιο ε, και θα αντιμετωπίσουμε ανταγωνισμό από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για επενδύσεις, αλλά και για την προσέλκυση ε, των ε, καλύτερων εργαζομένων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καλύτερο ε, περιβάλλον για τις επιχειρήσεις είναι όλα αυτά σημαντικά, αλλά η εκπαίδευση πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια που απαιτείται στην εκπαίδευση και να μπορέσουμε να συγχωνεύσουμε ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λόγω Τη εξωτερική μετανάστευση που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα δυστυχώ, την εσωτερική ε, μετανάστευση ω πρόβλημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη να χάνουν, ε, κάθε, να χρόνο εκατομμύρια εργαζόμενους ε, στι δυτικέ χώρε, αυτοί δηλαδή που θα χρειαζόντουσαν περισσότερο από όλου προκειμένου να ανοικοδομήσουμε τι χώρε μα. Να σα πω κάτι για την σύγκληση. Δεν υπάρχει διαρθρωτική σύγκληση χωρίς σημαντικότατες, σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις, αλλά χρειάζεται και πολιτική συνοχή και χρειάζεται χρηματοδότηση, αξιοποίηση των ταμείων της συνοχής, διευκολύνοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες και εξασφαλίζοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Πιστεύω ότι δεν ε, ωφελούνται μόνο οι καθαροί συνεισφέροντες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Όλα τα κράτη-μέλη ε, ωφελούνται από τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση και τα ταμεία. Αλλά πιστεύω επίσης ότι πρέπει να υπάρχει και να υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα για τους συνεισφέροντες ε, και να μην εξαρτούνται οι επενδύσεις μόνο από την συγχρηματοδότηση από τα ταμεία. Γι' αυτό και ε, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός ε, ο οποίος θα είναι ενταγμένος στην ΟΝΕ και που θα βοηθά στην παρακολούθηση των επενδύσεων και της χρηματοδότησης. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όλα τα ταμεία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα είναι πολύ πιο δύσκολο να κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κακά και να προσπαθούν διάφοροι κύκλοι να ωφελούνται και να πιστώνονται όλα τα καλά. Χρειάζεται εμπιστοσύνη. Τέλος, να πω κάποια λόγια από κροατική σκοπιά ως ε, νεότερης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από μια πολύ εξαντλητική ε, ύφεση την οποία ε, περάσαμε, Περάσαμε πλέον στην ανάκαμψη τα τελευταία δύο χρόνια και την ε, μείωση των, ε, του δημόσιου χρέους. Υπάρχει βελτίωση των ε, δικτών στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και αυτό έχει οδηγηθεί κυρίως από, την, από τις εξαγωγές και τις υπηρεσίες, χάρη στην συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πλέον χρειάζεται ο δημόσιος τομέας να περάσει από γρήγορες και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, ιδίω αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας για ένταξη στην ΟΝΕ, που είναι ένας από τους βασικότερους μας στόχους. Και σε αυτό χρειάζονται εθνικές μεταρρυθμίσεις, προετοιμασία σε εθνικό επίπεδο και το, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ακριβώς έχει αποδείξει ότι μπορεί να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία. Χωρίς συνεχείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ούτε η χώρα μου μπορεί να συγκλίνει με τις ε, ανεπτυγμένες χώρες, ούτε θα μπορέσει ε, η Ένωση στο σύνολό της να διατηρήσει την ηγετική της θέση, την ανάπτυξη και την ευημερία για τους πολίτες της. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε σήμερα. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Μιλόσεβιτς. Φυσικά γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές συνθήκες σε κάθε χώρα ε, είναι διαφορετικές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φάμπιαν Κέλλερ, Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υπηθέσεων της ε, Γαλλικής Γερουσίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι, ε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Επίτροπο, τους δύο Ευρωβουλευτές, ε, τον εκπρόσωπο του Κροατικού Κοινοβουλίου για τις παρεμβάσεις τους και να πω ότι και εγώ με τη σειρά μου θα σας παρουσιάσω την άποψη ενός εθνικού βουλευτή. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι χαίρομαι για αυτές τις ανταλλαγές μεταξύ εκπροσώπων των κοινοβουλίων, διότι αποτελούν ε, το κομβικό σημείο της ευάθυνσης ε, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Εγώ εκπροσωπώ τη Γερουσία στη Γαλλία, τη δεύτερη βουλή, και η Γερουσία... Ε, ε χρησιμοποίησε πολύ γρήγορα το νέο εργαλείο συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και γι' αυτό και ε, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων ε, ε, βάσει και του νόμου προγραμματισμού των δημοσίων οικονομικών από το 2011 το πρόγραμμα σταθερότητας εξετάζεται από το Κοινοβούλιο μας πριν το διαβιβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θεωρώ ότι αυτό αντανακλά την δημοκρατική απέτηση και την εξοικείωση με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε καμία οικονομική παρέμβαση χωρίς ε, την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο καθένας από εμά εξασφαλίζει την ομοποίηση και την πρόσβαση σε δύσκολες ορισμένες φορές απεφάσεις. Ε, ή αντιστρόφως, οι βουλευτές μας είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βάλουν την ευρωπαϊκή πτυχή στις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι από το 2010 και μετά είχαμε πολύ σημαντικές πρόοδους. Αυτό ε, είναι αποτέλεσμα μιας ευρωπαϊκής ε, πρωτοβουλίας που ξεκινήσαμε μαζί με τον συνάδελφό μου στη Γερουσία επιμείναμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό εξάμεινο και συμβάλλει πολύ και εδώ θα ήθελα να εκφράσω και μία ευχή, την εξέφρασα και πέρσι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω την ε, αποτελεσματικότητα αυτών των διακοινοβουλευτικών ε, συνεδριάσεων θα πρέπει να υπάρχουν συμπεράσματα ή ψηφίσματα τα οποία θα μπορούσαν από εκεί και πέρα να επισυμποποιηθούν και να διαβιβάζονται στα διάφορα ε, όργανα λήψης αποφάσεων. Να έρθω τώρα στις προτεραιότητες που επιβάλλονται για το 2018. Η οικονομική ανάκαμψη υπάρχει μεν, αλλά πολλά κράτη-μέλη την αμφισβητούν. Υπάρχει ποσοστό της ανεργίας αρκετά υψηλό, ε, ιδίως για τους νέους, ε, όπως ανέφερε προηγουμένως ε, και ο συνάδελφος. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και η οικονομική ανάκαμψη φυσικά ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και επανεξισορρόπηση των μακροοικονομικών πολιτικών και η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει ε, μία ε, σταδιακή εξομάλυνση των διαδικασιών της. Πρέπει να κινητοποιήσουμε βέβαια και άλλα μέσα, καταρχάς να εφαρμόσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές στήριξης των επενδύσεων. Υποχρονόμαστε βεβαίως διότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συντονισμού, να συντονιστούν και αυτή είναι και η έννοια, κύριε Επίτροπε, των αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, να έχουμε ε, ε, μια εξισορρόπηση της μακροοικονομικής κατάστασης. Για τη Γαλλία αυτό μεταφράζεται στις απαραίτητες προσπάθειες για να σεβαστούμε τα κριτήρια του δημόσιου ελλείμματος, τα οποία επιβάλλονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έγιναν προσπάθειες από τη χώρα μας και ο στόχος αυτός ε, αποτέλεσε και ε, το βασικό στοιχείο που λάμβανε υπόψη του ο υπουργό ε, Οικονομικών, όπως ανέφερε και στη Γερουσία σε ομιλία του πρόσφατα. Το 2016 προτάθηκε η έξοδος της Γαλλίας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. Θα εφαρμοστεί την επόμενη άνοιξη και ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει ε, πρόβλημα, αλλά φυσικά θα πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Ε, μόνο σεβόμενοι τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει θα καταφέρουμε στην πραγματικότητα να έχουμε συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών ε, και θεωρώ ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να κινητοποιηθούν όλα τα κράτη-μέλη για να έχουμε μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική στο όνομα της σταθερότητας, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα υπάρχουν ε, και εκλογές, ε, το, είχαμε και εκλογές το 2017 για τη Γαλλία και το 2018 είναι η χρονιά που θα συζητηθούν πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη η Τραπεζική Ένωση, την οποία θα συζητήσουμε και αργότερα, αλλά και η εμβάθυνση της Ένωσης των Κεφαλαγορών. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται στην ενιαία αγορά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να ανανεώσουμε τα εθνικά φορολογικά μας συστήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ε, ε, ανάγκη και την αυξανόμενη ε, δράση της ψηφιακής οικονομίας και την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Προηγουμένως ακούσαμε πόσο σημαντική είναι αυτή η καταπολέμηση. Επίση, την ενιαία φορολογική βάση επιχειρήσεων ε, θα πρέπει ε, να υπάρχει και ε, βούληση και από τις επιχειρήσεις για να το εφαρμόσουμε αυτά. Να χαιρετήσω τα όσα κάνουν ο κύριος Λαμασούρ και η Περβάνς Περές για να μπορέσει να ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό και επίσης να πω ότι ελπίζω σε μία από τι επόμενε συναντήσει μα να μπορέσουμε να αποφασίσουμε όλοι μαζί ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό, διότι οι πολίτες περιμένουν. Οι Υπουργοί Οικονομικών είχαν ε, χαιρετήσει το 2016 την έναρξη αυτού του προγράμματο. έγιναν κάποιε προτάσει βελτίωση, για παράδειγμα για να ληφθεί υπόψη και υποστήριξη στην έρευνα. Τέλος, ε, η Γαλλική Γερουσία προσπαθεί να κινητοποιηθεί για την ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη φοροαποφυγή. Ε, αρκετές προσπάθειες για την ψηφιακή ε, φορολόγηση, διότι υπάρχουν ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικών εσόδων που χάνονται λόγω απάτης στο διαδίκτυο και οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι δίκαιο το σύστημα για όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρωτοβουλίες αυτές για τα θέματα αυτά δεν μπορούν να είναι αμυγός εθνικές. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κοινοβουλίων για να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε μορφή φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να προσαρμογράψουμε αυτή την ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές μας. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα των Επιτροπών που διοργανώνουν τη σημερινή διάσκεψη να καλωσορίσω όλους τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια Έχουμε 133 συμμετέχοντες σήμερα, είναι ρεκόρ ο αριθμό αυτός για τη συμμετοχή. Νομίζω λοιπόν ότι η διάσκεψη αυτή ε, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία και χαιρετίζω το στοιχείο αυτό καθώς και τις πολύ καλές ε, παρεμβάσεις που είχαμε μέχρι στιγμής από τους ομιλητές μας. Και τώρα πια ε, ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Πρώτος ομιλητής είναι η κυρία Ροντρίγκε από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Τρία λεπτά υπενθυμίζω ο χρόνος αγόρευσης και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε εδώ. Θα μιλήσω ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ε, κοινωνικό πυλώνα. Παρατήρησα ότι οι περισσότεροι ομιλητέ τόνισαν το γεγονό ότι αυξάνονται οι, Ευρωπα... οι ανισότητε, οι κοινωνικέ ανισότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τι προσπάθειε που έχουν γίνει για την καταπολέμησή του. Και ο κοινωνικό πυλώνα είναι πράγματι μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία προκειμένου να δοθεί απάντηση στις κοινωνικές ανισότητες, νέους παιδιά, άνδρες και γυναίκες, την ενίσχυση των προδιαγραφών, τη βελτίωση των προδιαγραφών και την αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών ανισοτήτων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όποια δουλειά και να έχει κανείς, θα πρέπει ο μισθός να εξασφαλίζει, να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και κοινωνική προστασία. Και αυτή είναι, ε, αυτή είναι μία από τις βασικές υποσχέσεις αυτού του κοινωνικού πυλώνα. Ταυτόχρονα θέλουμε όμως να υπάρχει και σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της Ευρώπης προκειμένου να παρέχονται ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντική η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί πράγματι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρέπει να υλοποιείται ως μια μεγάλη διαδικασία για την σύγκληση προς τα πάνω, οικονομικά και κοινωνικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει σημαντικές προτάσεις. Έχουμε πλέον δίκτες για τη μέτρηση αυτής της σύγκλησης. Η μεγάλη δοκιμασία όμως θα έρθει όταν ε, θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες όπως το κάνουμε με τις, κοινωνικές, με τις οικονομικές ανισότητες. Και γι' αυτό το σκοπό χρειαζόμαστε βεβαίω μεταρρυθμίσεις αλλά και επενδύσεις. Και για να έχουμε επενδύσεις πρέπει να πάμε παραπέρα όσον αφορά τις ε, οικονομικές και επενδυτικέ μας ικανότητες, να αξιοποιήσουμε όλα τα, όλους τους πόρους που έχουμε, ιδιωτικούς και δημόσιου, τα δημοσιονομικά εργαλεία που έχουμε, το πολυετές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και τέλος πρέπει να εξοπλίσουμε την νομισματική μας ζώνη με δημοσιονομικές ικανότητε Αυτή είναι η όρη προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική κοινωνική αλλά και οικονομική σύγκληση. Ευχαριστούμε. 30 ε, δευτερόλεπτα λιγότερα από όσα σου είχα δώσει. Επόμενος ομιλητής. Ο Γιάννης Φούκανς από το Λιτωνικό Κοινοβούλιο, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Γενικά η χώρα μου, η Λετωνία, χαιρετίζει και υποδέχεται ε, με χαρά τις ε, κατευθυντήρες γραμμές που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ε, για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πρέπει να συνεχίσουν το έργο για τη διευκόλυνση των υπονδύσεων, την ε, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η πρόοδος όμως είναι ε, άνηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναγνωρίζεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική έκθεση για την ανάπτυξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ιδίω στο τομεί όπου έχουμε μείνει πίσω. Η, η ανάγκη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς έχουμε θέσει το στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Γενικά η Λετωνία συμφωνεί με τις συστάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να τονίσουμε τον, τον ρόλο που ε, θα κληθεί να διαδραματίσει και η ενιαία αγορά, ιδίως η ψηφιακή ενιαία αγορά. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ενιαία αγορά και να καταργηθούν όλα τα εμπόδια στην κίνηση ε, προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων και κεφαλαίων. Και για το σκοπό αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί και η εσωτερική κινητικότητα στην αγορά εργασίας ε, και να σταματήσει ε, η μονομερής ροή από τις φτωχότερες προς τις πιο πλούσιες χώρες εργαζομένων. Είναι σημαντικό επίσης να, να ενισχυθεί η ΟΝΕ και η Λετωνία υποστηρίζει την, το σχέδιο δράσης για την ενοποίηση των κεφάλαιων αγορών. Χρειάζεται να υπάρξει ανάπτυξη των κεφαλαίων αγορών σε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταβληθούν ε, προσπάθειες και στον τομέα της καινοτομίας. Στις 6 ε, Νοεμβρίου του 2017 οι Υπουργοί Οικονομικών των τριών βαλτικών χωρών υπέγραψαν ένα μνημόνιο ε, αλληλοκατανόησης για την ανάπτυξη της περιφερειακής κεφαλαίου στη Βαλτική. Εκεί τονίζεται η δέσμευση και η προσήλυση των ε, τριών βαλτικών χωρών στην ανάπτυξη μιας ενιαίας κεφαλαίου με συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το σχετικό νομικό πλαίσιο, η εισαγωγή νέων νομικών εργαλείων και η δημιουργία των ε, απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία αυτής της κεφαλαίου αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής. Σάουρα Πέντρο. Από την Ισπανία, από το Κογκρέσιο της Ισπανίας, σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύντομα, κάποιες ιδέες θέλω να σας μεταφέρω, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η πρώτη μου ιδέα, λοιπόν, είναι ότι σε σχέση με αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο, πιστεύουμε ότι τα σχέδια μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων και τα σχέδια σύγκλησης πρέπει να περιλαμβάνουν δίκτες. Δηλαδή να συμπεριλάβουμε και δίκτες καλής διακυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα βοηθούσε να πετύχουμε τη σύγκληση αυτή τη δημοσιονομική που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πιστεύουμε ότι θα έπρεπε οι συζητήσεις που γίνονται στα εθνικά κοινοβούλια να φτάνουν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερώνονται για αυτές τις συζητήσεις, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν φτάνει η στιγμή της υλοποίησης. Η τρίτη ιδέα είναι ο, ο επαναπροσανατολισμός του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Οι κανόνες δηλαδή που ισχύουν στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μιλάω για συγκεκριμένους στόχους αξιόπιστους που θα βάλουμε μέσω πρόθεσμα με μια πιο απλή λογιστική που θα βοηθήσει και την ευελιξία των δημοσιονομικών κανόνων ε, καθορίζοντας ε, ανεξάρτητες αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι απόλυτα συμβατό με τη λογοδοσία, με περισσότερη δημοκρατία και με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Και τέλος, η τελευταία μου ιδέα που θέλω να σας μεταφέρω εδώ, σε εσά, του συναδέρφους μου ευρωβουλευτές ή βουλευτές από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι εξή. Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για να δημιουργηθούν πραγματικές ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτός είναι ένας σωστός δρόμος και αποτελεσματικός δρόμος για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Τζον Λέιχαρτ. Ιρλανδία και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Είναι δύο θέματα που θέλω να θίξω εδώ. Το ένα είναι τα μίξη που να δάνεια, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε η Επίτροπος. Η κατάσταση στην Ιρλανδία είναι ότι έχουμε 20.000 υποθήκες περίπου, που βρίσκονται σε πίεση και πρέπει να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα ή κάτι να γίνει με αυτές. Υπάρχουν όμως τα λεγόμενα ε, voucher funds που αγοράζουν τέτοιες υποθήκες σε πολύ χαμηλές τιμές, με μεγάλη έκπτωση. Και αυτή η έκπτωση δεν προσφέρεται όμως στους ιδιώτες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Γιατί αυτά τα voucher funds δεν είναι κανονικά, δεν είναι επίσημα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να συζητήσουν με τους πελάτες τους για να υπάρξει εξυπηρέτηση αυτών των δανείων, αντί να πουλάνε πακέτα τέτοιων υποθηκών και τέτοιων μη εξυπηρετούμενων δανείων στα Vulture Funds αν θέλουμε μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη, αν μη τι άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε δάνειο υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό που έχουν σχέση και με επιχειρήσει. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν οι άνθρωποι αναγκάζονται να χάσουν τα σπίτια τους. Και αυτό επιβαρύνει επιπλέον το κράτος. Και μερικές φορές έχουν αυτοκτονήσει και άνθρωποι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση από τις τράπεζες. Αυτό ήταν το πρώτο μου θέμα. Το δεύτερο είναι ε, για το σύστημα τραπεζικών εγγύσεων, που αποτελεί ένα πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης. Η πρόοδος έχει σταματήσει τελευταία, δεν ξέρω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας ενημερώσει πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πάντως για το πρώτο μου θέμα, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να αποθαρρύνουμε τις τράπεζες να πουλάνε τις υποθήκες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε αυτά τα ε, ταμεία, τα μη επίσημα, γιατί πίσω από κάθε δάνειο βρίσκεται μια ζωή. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε. Όπως ξέρετε, οι πιέσει από τον νέο επόπτη πηγαίνουν προ την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που επισημάνατε, που ελπίζετε μάλλον. Πρόκειται για ένα θέμα όμως το οποίο γνωρίζουμε. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα μέτρα στον τομέα αυτό. Τώρα από την Ισπανική Γερουσία, από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Μαραγκούλο. Η κυρία, συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις κοινέ προτεραιότητες ε, στις οποίες αναφερθήκατε όλοι νομίζω ε, και στις οποίες είμαστε βυθισμένοι όλοι στην Ισπανία. Αναφερόμαστε σε ανταγωνιστικότητα, σε κατάρτιση, κοινωνικό θεματολόγιο, καθώς επίσης και την ανάγκη αντιμετώπισης αρκετών ε, σημαντικών προκλήσεων, όπως είναι η δημογραφική πρόκληση και το τι προϋποθέτει ε, η προώθηση της απαραίτητης της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και στις χώρες μας, όπως κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διαπιστώσαμε και σήμερα αναφερόμαστε σε μια οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ισπανία έχουμε οικονομική ανάπτυξη πράγματι ε, και αντίθετο από ότι σε άλλες περιπτώσεις όπου αναφερόμαστε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, τώρα ε, πρέπει να αναφερθούμε στην αποδεδειγμένη δυνατότητα των μεταρρυθμίσεων να βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. και εδώ θα ήθελα να τονίσω στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μου, όπου για τέταρτη συναπτή χρονιά έχουμε σημαντική ανάπτυξη και υπάρχει και ένα ποσοστό ανάπτυξης για το 2017 3,1% και δημιουργούνται και θέσεις απασχόλησης. Αναφερόμαστε λοιπόν σε κοινέ προτεραιότητες ε, και το θεματολόγιο, όπως και σε άλλες ε, κυβερνήσεις, επικεντρώμαστε ε, στην κατάρτιση, σε πολιτικές για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε απασχόληση και σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ψηφιοποίηση, η ψηφιακή ε, ανάπτυξη και αναφέρθηκε και στο Προεδρείο και πρέπει να πω ότι αναφερθήκε και στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών της Ισπανίας και συστήθηκε μια ομάδα εργασίας για να δούμε τα μέσα και τα μέτρα τα οποία ε, εφαρμόζονται, να υπάρχει συντονισμός μεταξύ εννέα Υπουργείων και να έχουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η ψηφιακή αυτή ανάπτυξη να βοηθήσει ως εργαλείο και να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά ταυτόχρονα και η ψηφιοποίηση ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ε, διαφυγή και κοινωνική συνοχή, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποτελεί πηγή αύξηση ευκαιριών, ε, εγγύηση ισότητα ευκαιριών σε περιοχέ τις οποίε υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες ε, λόγω εγκατάλειψη από πλευρά του πληθυσμού ή πιο αεροκατοικημένων περιοχών και ε, στην υπηρεσία αυτή τη κοινωνική συνοχή. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη και οι μεταβλητές που παρακόλλησαν την ανάπτυξη ήταν η ανεργία και οι δημογραφικές προκλήσεις και πιστεύω ότι οι διαδικασίες δημιουργίας νέων ε, ψηφιακών εργαλείων και προκλήσεις όπως η ε, διασύνδεση των διαφόρων περιοχών και ε, η εκμετάλλευση των συνεργειών που δημιουργούνται είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτό θα ήθελα και αυτό μου άρεσε από όλες τις παρεμβάσεις που άκουσα και πιστεύω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γκαμπριέλα Κρέτσου από την Ρουμανική Γερουσία τώρα, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να επιστήσω για άλλη μια φορά την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουμε πρόβλημα διάγνωσης. Οι λανθασμένοι δείκτες ε, μας δίνουν μια λιγότερο ρεαλιστική εικόνα της κοινωνίας και ε, οδηγούν σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι κατάλληλες. Αυτή τη στιγμή η βασική μακροοικονομική έλλειψη ισορροπίας βασίζεται ε, στο δίκτυο ε, εισόδημα εργασίας, κεφαλαϊκό εισόδημα και υπάρχει πρόβλημα κατανομής. Και αυτό δεν είναι μόνο κοινωνικό θέμα, αριστερά κόμματα και συνδικάτα τα οποία θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, αλλά αντανακλάται και στις στον ακατάλληλο δίκτυ επενδύσεων κατανάλωσης που είναι ο βασικός ε, ε, δείκτης για να μετρέσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η ανισορροπία είναι παγκόσμια και το γεγονός ότι εξάγονται οι αρνητικές της συνέπειες ε, για την κοινωνία μας δεν είναι πλέον δυνατόν. Θα πρέπει να δούμε τους 14 δείκτες που εξελογούν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες είτε στις εκθέσεις αναχώρα εντός ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είτε οπουδήποτε αλλού. Δεύτερον, έχουμε μια οικονομία χωρίς σύνορα που αποκαλείται μια αγορά και θεωρείται ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τούδε. Αλλά ε, έχουμε δείκτες με σύνορα, εθνικούς δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση πολιτικών και την αξιολόγηση της υλοποίησής τους για τη γενικότερη ε, σύγκληση που θα χρειαστούμε για να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης ο οποίος ε, χρησιμοποιείται είναι ο δείκτης ε, του κατακεφαλήνα ΑΕΠ και την αγοραστικής αξίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όμως αν θέλουμε να μειώσουμε τα ποσοστά της ανάπτυξης και κυρίως τα κενά σε δυνατότητες ανάπτυξης. Το ΑΕΠ καταδεικνύει τι συμβαίνει σε μια χώρα όχι τι παραμένει σε αυτή τη χώρα. Και πρόσφατα αποδείχθηκε ότι οι επιστροφές και ο επαναπετρισμός των εσόδων είναι υψηλότερους από τα ε, κονδύλια τα οποία μπαίνουν ε, στα δημόσια ταμεία, δηλαδή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μείων της συμβολής στον Ευρωπαϊκό Κορβανά για όλες ε, τις πολιτικές στις οποίες ανήκει η χώρα μου η Ρουμανία. Οι δείκτες αυτοί λοιπόν είναι παραπλανητικοί διότι ε, επικεντρώνονται στο παρόν και δεν ε, λαμβάνουν υπόψη τους και το αποθεματικό που είναι ο πλούτος μιας κοινωνία και ε, η πρόβλεψη για τις δυνατότητες ανάπτυξή της. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη συνδέεται με τον πλούτο και με το ανθρώπινο κεφάλαιο και λιγότερο με το ΑΕΠ και το ποσοστό του ΑΕΠ. Αν ε, λοιπόν δούμε τα εισοδήματα, βλέπουμε μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η σύγκληση των κερδών είναι εξαιρετική. Στη χώρα μου είναι πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Το ε, εισόδημα των οικοκυριών όμως από την άλλη είναι στο 32% περίπου. Η ανάπτυξή μας λοιπόν έχει πάει προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και δεν υπάρχει καμία σύγκληση, υπάρχει απόκληση. Αν δούμε και τις αποκλήσεις λόγω του ευρώ, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οι ανισότητες εντός κάθε κράτους μέλους και μεταξύ κρατών μελών αποτελούν το βασικό στόχο των ευρωπαϊκών πολιτικών και των συντονισμένων ε, εθνικών πολιτικών, ε, όπως ε, πολλοί από εσάς επισημάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε που μας ε, υπενθυμίσατε την, την ανεπαρκή θέση ή προσοχή που έχει δοθεί στις επενδύσεις. Η Μαργαρίτα Μάρκες έχει τώρα το λόγο από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο και τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές που ξεκίνησαν αυτήν την συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές αυτής της ε, διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψης. Η Επίτροπος Τάισεν υπενθύμησε ένα στοιχείο που βεβαίως το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Υπάρχει λοιπόν οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο οι ανισότητες παραμένουν σημαντικότατες και εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας απευθύνω. Χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή όσον αφορά τον οικονομικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Κατά τη γνώμη σας. Υπάρχουν επαρκείς πολιτικές για την σύγκληση. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Αφενός λοιπόν η οικονομική ανάπτυξη και οι κοινωνικές ανισότητες που ταυτόχρονα αυξάνονται. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και τα δύο. Θα ήθελα να, κάνω κάποιες, να με κάνω μια τοποθέτηση σε σχέση με τις συστάσεις αναχώρα. Νομίζω βασικό ε, στοιχείο είναι η ενεργή συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το να διαβάζονται απλώς κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη Ε, τα οποία μάλιστα καλούνται να απαντήσουν μέσα σε δύο-τρει μέρε, δεν αρκεί. Οι συστάσει αυτέ πρέπει να είναι αποτελεσματικέ και με δεδομένε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να υπάρχει ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των κρατών μελών στην κατάρτιση αυτών των συστάσεων. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να θέσω αφορά τον κοινωνικό πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει να σα πω ότι με χαρά μου άκουσα τη Μαριάν να λέει ότι έχει δημιουργηθεί ένα βαθμολόγιο το οποίο πλέον θα συμπεριλαμβάνεται και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ταυτόχρονα όμως ε, έχω την άποψη ότι είναι πολύ δύσκολο οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες να κατανοήσουν ότι υπάρχουν στόχοι για δημοσιονομικά ζητήματα αλλά όχι για κοινωνικές υποθέσεις ή κοινωνικές πολιτικές. Αυτό το βαθμολόγιο λοιπόν θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όμως δεν μπορεί να είναι απλώς μια συμβολική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πραγματικές δράσεις από την πλευρά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και τέλος, θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση της Φάμπιαν Κάλερ που είπε ότι θα πρέπει στο τέλος αυτών των συναντήσεων να υπάρχουν ψηφίσματα και συγκεκριμένες προτάσεις. Η Βάνα Μαλέτης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Τονίσατε όλοι το γεγονός ότι υπάρχει ανάπτυξη πλέον, χωρίς όμως να είμαστε υπερενθουσιώδεις, γιατί δεν έχει αντικατοπτρεστεί στην καθημερινή ε, ζωή των πολιτών. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την βελτίωση των μισθών, την αύξηση των μισθών και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο και το φάσμα της φτώχειας και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε ε, τρόπο ε, αποτελεσματικότερο για τη χρηματοδότηση και την ε, ιεράρχηση των επενδύσεων. Τι ακριβώς τελικά χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της καινοτομίας και των διαδικασιών μεταρρύθμισης και μεταμόρφωσης της οικονομίας. Το Ταμείο Juncker Στρατηγικών Επενδύσεων ε, εξυπηρετεί τον στόχο της χρηματοδότησης ε, δημόσιων και ιδιωτικών έργων, την, την συγχώνευση και τον συνδυασμό ε, ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων σε συγκεκριμένα έργα, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ανοίξουμε περαιτέρω την χρηματοδότηση για να μπορέσει να ενισχυθεί η καινοτομία, να χρηματοδοτηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις και στη συνέχεια να τους δοθεί η δυνατότητα να περάσουν στο επόμενο στάδιο, από startup να γίνουν scale-up, γιατί όλα αυτά τα μέτρα θα σημάνουν σημαντικές και πραγματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Ευχαριστώ. η κυρία Φόλκανας Κίσνερ από τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου και τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μας ικανοποίηση ε, βλέπουμε και διαπιστώνουμε και εμείς την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και ελπίζουμε πράγματι αυτή να είναι η ανάπτυξη, η ανάκαμψη να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ε, με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τους ομιλητές που τόνισαν την ανάγκη που υπάρχει να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή, να αντιμετωπιστούν οι διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες κτλ. Ταυτόχρονα όμως και την ανάγκη να βελτιωθεί η ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αξιοποιηθούν τα ωφέλη που μπορούν να προέλθουν από την κοινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη κτλ. Ακούγοντας λοιπόν τα σχόλια που ακούστηκαν, ε, κάτι που ε, έπεσε στην αντίληψή μου είναι η αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικότητας και των φιλοδοξιών που εκφράστηκαν και ε, θυμήθηκα μια ομιλία της κυρίας Μέρκελ εν ώψη των στόχων του 2030 όπου ανέφερε ότι η Ευρώπη ε, ε, αντικατοπτρίζει το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περιλαμβάνει το 50% των, των παγκόσμιων κοινωνικών δαπανών θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη μας γιατί δεν γίνεται ταυτόχρονα να υπάρχει ε, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και κοινοτομίας που χρειαζόμαστε με την τέταρτη βιομηχανική ε, επανάσταση, τη ρομποτική και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα έρθουν ε, στις κοινωνίες μας τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα να επιμένεις ότι πρέπει να συνεχίσει η εκθετική αύξηση των κοινωνικών δικτύων, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής. Είναι, ένα σκέψη, είναι μια σκέψη ε, την οποία θα ήθελα να καλέσω τους ομιλητές να εξετάσουν και εκείνοι και αν μπορούν να τοποθετηθούν. Ευχαριστούμε. Αντρέσκουν και τώρα, γερμανικό Bundesbank από την Δερλίνγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές που αναφέρθηκαν στο ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας με τέτοιο σθένος, διότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό που παρακολουθούμε σε διεθνές επίπεδο είναι ότι ολοένα και περισσότερο υπάρχει μια αλλαγή του προτύπου. Ε, πολλοί διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΩΣΑ, ε, η Ευρωζώνη έτσι κι αλλιώ, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακόμα και το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο ε, ασχολούνται και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της κοινωνικής ανισότητας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ε, αναφέρθηκε και η συνάδελφος από τη Ρουμανία για παράδειγμα ότι οι ανισότητες αυτές δεν αποτελούν κριτήριο του βαθμολογίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όχι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του κοινωνικού πυλώνα. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτός ο κοινωνικός πυλώνας δεν θα είναι αρκετάς για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω το ερώτημα στην Επίτροπο Τάισεν, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε. Δεύτερον, υπάρχει μακροοικονομική, οικονομική ανισομετρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ε, ε, επαναλήφθηκε και το στοιχείο ε, ότι το η Γερμανία ξεπερνά το όριο του 6% πλεονάσματος για άλλη μια χρονιά φέτος. Πια 8,1 είναι το επίπεδο στο οποίο κινείται αυτή τη στιγμή φέτος. Τι μέτρα θα πάρετε για να περιορίσετε αυτό το πλεονάσμα. Αυτό είναι αρνητικό ακόμα και για το γερμανικό λαό γιατί σημαίνει ακριβώς ότι η μισθή ε, είναι πάρα πολύ χαμηλή, ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κοινωνικές ε, δαπάνες και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στην ε, φορολογική εναρμόνιση. Είπατε κι εσείς όλοι οι ομιλητές ότι πράγματι οι διαφορές μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών αποτελούν πρόβλημα ακριβώς γιατί δίνεται η δυνατότητα σε μεγάλους διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους να επιλέγουν πού ακριβώς θα φορολογήσουν τα κέρδη τους. Ε, θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια κοινή ενιαία φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώς για να αρθούν αυτά τα εμπόδια και τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη φορολογία. Ο Τζανπάιλο Γκάλι από τη ε, Βουλή ε, των, ε, της Ιταλίας, από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλες οι παρατηρήσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα λένε ότι ωραία υπάρχει ανάκαμψη στην Ευρώπη, όμως σε πολλές χώρες ο κόσμος δεν έχει αισθανθεί ακόμα αυτά τα ωφέλη ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ μερικός θα έχει αισθανθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη σε αυτό που είπαμε, ότι υπάρχουν ανισότητες. Εν μέρη μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος ώστε η εν παση περιπτωσει πολυ μερικο αυτή να γίνει αισθητή. Έχουμε να οφειλεται στο γεγονο εκατομμύρια φτωχών, εκατομμύρια ανέργων και πράγματι οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες βρισκόνται χρωμένες σε μεγάλο βαθμό. Κάτι που έχει επιπτώσεις στην μακροοικονομική μας πολιτική και όσον αφορά τις ειδικές συστάσεις χώρα που θα δούμε σε μερικές εβδομάδες, αυτό θα γίνει ακόμα πιο αισθητό. Ιδίω θέλω να αναφερθώ εδώ τώρα στην πολιτική προπολογισμού, κάτι το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συγκεκριμένα έχει βοηθήσει χώρες να κατευθύνουν τον προϋπολογισμό τους έτσι ώστε να μειωθεί το χρέος τους. Κυρίως οι χώρες που έχουν ιδιαίτερα υψηλό χρέος. Όμως είναι ζωτική σημασία να γίνει μια στάθμιση ε, στις συστάσεις αυτές προσπαθώντας να βρούμε ε, το σωστό ρυθμό της φορολογικής εξυγένωσης. Αν δεν βρούμε τη σωστή ταχύτητα, το σωστό ρυθμό, τότε κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε σύγκρουση και σε ζημιά. Οι στόχοι που θα καθοριστούν πρέπει να γίνονται κατανοητοί, να είναι αξιόπιστοι και οι εθνικές αρχές και το εκλογικό σώμα να κρίνουν ως κάτι το αξιόπιστο. Πρέπει δηλαδή οι στόχοι να είναι στόχοι ρεαλιστικοί που να μην αλλάζουν κάθε χρόνο ή ακόμα και δύο φορές το χρόνο. Εγώ διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλεξ Μπόντρι. Λουξεμβούργο, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρο, όπως κι άλλοι, έτσι και εγώ θέλω εδώ να χαιρετήσω τα τελευταία στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την ανάπτυξη που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη επανέρχεται στην ανάπτυξη παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ανισότητες κοινωνικές μεταξύ των χωρών μελών, αλλά ακόμα και στην ίδια χώρα. Οπότε, ναι, μεν εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που αυτός ο κοινωνικός ο πυλώνας θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό βαθμολόγιο, αλλά το βαθμολόγιο αυτό και αυτή η μικρή κοινωνική διάσταση στην οικονομική διακυβέρνηση παραμένει ξένο σώμα μέσα σε ένα σύστημα που έχει προκαθοριστεί αποκλειστικά ουσιαστικά για την οικονομία, για τα δημοσιονομικά. Οπότε θέλω να ρωτήσω την Επίτροπο Τέσσερ το εξή. Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι αυτή η κοινωνική διάσταση δεν θα παραμείνει ο φτωχό συγκινής, αλλά ότι θα υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι για την δημοσιονομική ισορροπία και την ισορροπία των δημοσιονομικών των χωρών μελών. Και αν λάβουμε υπόψη μας αυτό που είναι αναγκαίο, δηλαδή η ισότητα, πώς θα τηρηθεί αν τηρήσουμε και τη δημοσιονομική ισορροπία. Γιατί αν δράσουμε στις κοινωνικές ισορροπίες, δηλαδή προσπαθήσουμε να πετύχουμε κοινωνική ισορροπία, αυτό θα κοστίσει χρήματα. Οπότε πώς θα συμβιβάσουμε τη δράση μας στον κοινωνικό τομέα και συγχρόνως θα τηρήσουμε τους κανόνες σταθερότητας και ανάπτυξης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει αύξηση μισθών και αγοραστική δύναμη. Κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου στο Λουξεμβούργο για την τιμαριθμική προσαρμογή. Πώς όλα αυτά θα συνδυαστούν όμως με τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι να υπάρξει προσαρμογή της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Ευχαριστούμε. Τη τώρα. Ε, Πολωνική Γερουσία. ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η μετανάστευση, που είναι η άμυνα και η καινοτομία. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν άλλα, αλλά θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια γενικότερης πολιτικής και γενικότερων πολιτικών που οδηγούν στις ανισότητες. Ο κύριος ε, Χάρτμαν αναφέρθηκε έμεσα σε αυτά όταν μίλησε για τις ανισότητες που υπάρχουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επίρου, αλλά και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και περιφερειακό. Η οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση των ανισοτήτων. Η δικιά μας, η αντιπροσωπεία και η Πολωνία, θα ήθελα να υπάρχει κάποια συνέπεια. Είπατε ότι όταν ο καιρός είναι καλός, τότε φτιάχνει κανείς τη σκεπή του σπιτιού του. Εντάξει, αλλά δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και εμείς περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι συνεπής και να φροντίσει να πάψει να υπάρχει αυτή η ανισότητα. Η Πολωνία φυσικά και είναι διαθέσιμη να συζητήσει όλα αυτά τα θέματα και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και την πρόκληση του Brexit. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτή τη συζήτηση επίσης. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια που θα λείψουν, αυξάνοντας, ενδεχομένω τον προπολογισμό αλλιώ, αλλά δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Οπότε η έκκληση που κάνω είναι να επανέλθουμε στις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να... και τότε μόνο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής. Ε, με χαρά δίνω το λόγο σε ένα μέλος της Επιτροπή των Περιφερειών, την Όλγα Ζρίχαιμ, προσκεκλημένο μέλος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαρά μου να σας ξαναδώ εδώ σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα ως εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών να μπορώ να λάβω το λόγο. Ε, θεωρούμε ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης που ενδιαφέρονται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα πρέπει να συμμετέχουν, επομένως και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν και κάποιες εξουσίες και αρμοδιότητες ε, στις περισσότερες από τις πολιτικές που ενδιαφέρουν το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όλες οι συστάσεις αναχώρα το 2017 έχουν μια ιδιοφική διάσταση και μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίσουν ενεργό ρόλο ε, την 1η Φεβρουαρίου εγκρίθηκε στην ε, Επιτροπή των Περιφερών ένα ψήφισμα για την ε, ε, ανάπτυξη το 2018, για την ετήσια άκρηση ανάπτυξη και εδώ αναφερόμαστε στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, να σταματήσουν να υπάρχουν κόμματα για τι επενδύσει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι περιφέρειες να θεωρούνται εταίροι στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίση, θέλουμε να ενισχύσουμε και τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ για το 2030. Επιπλέον, το ψήφισμα επισημαίνει ότι η πολιτική των περιφερειών θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο που θα ε, ε χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εδαφική και κοινωνική συνεχή και να βασίζεται και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ε, δράτω με τις ευκαιρίες εδώ, ε, λόγω της συζήτησης για τις διάφορες πτυχές ε, της βελτίωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μια συζήτηση ιδιαίτερα δυναμικές, διότι οι συζητήσεις για την ε, νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η βάθηση της ΟΝΕ θα επιτρέψουν να δούμε και τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θεωρούμε ότι ενδιαφέρει και την πολιτική ε, συνοχής και το νέο μέσο χρηματοδότησης για να υποστηρίξουμε τι τις μεταρρυθμίσει. μεταρρυθμίσεις Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Η υλοποίηση των συστάσεων ονοχώρα δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για τι συστάσει αναχώρα όσον αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που δεν έχουν πραγματική ε, νομική βάση και α το αναγνωρίσουμε, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Και αυτά παρά τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσει τον αριθμό και να ε, επικεντρωθεί σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε ε, σε 12 ή 18 μήνε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για του οποίου δεν υλοποιούνται αυτέ ε, τεχνικές αρμοδιότητες, διοικητικές ε, δυνατότητες, φυσικά και χρηματοδότηση, αλλά και ε, ο αριθμός των εθνικών προβλημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τίποτα δεν μπορεί να αποζημιώσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πόροι σε εθνικό επίπεδο και ενωμένο, επομένως θα πρέπει οι συστάσεις αναχώρες εάν να θεωρούνται ε, δεσμευτικές θα πρέπει να απαντούν αντίστοιχα και τα κράτη-μέλη. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ως εταίροι και θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε να αυξάνεται η συμμετοχή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και επίσης ζητούμε η συμμετοχή αυτή να, ε, να ξεκινάει από την αρχή, από την κατάρτιση, από εκεί και πέρα στην υλοποίηση στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση. Προτείναμε και ένα κώδικα διοντολογία για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο, που διαιρείται σε δύο τμήματα. Μία ανάλυση των ευκαιριών σε ε, εδαφικό επίπεδο και επίση πώς μπορούν να συμμετέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχέ ως εταίροι στη σύλληψη και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ζητάμε λοιπόν αυτό, αλλά ζητάμε και την εταιρική σχέση. Μία ιδέα την οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2016, υποστηρίζοντας την ιδέα ενός κώδικα διοντολογία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ω ανάγκη να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέριψε την πρότασή μα για ένα κώδικα διοντολογία γιατί φοβήθηκε ότι δεν θα γίνει σεβαστή η αρχή τη επικουρικότητα. Αντιθέτω, πιστεύουμε ότι η επικουρικότητα θα ε, τηρηθεί εάν οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ λεμφθούν υπόψη στη διαδικασία, διότι αποτελούν ε, άμεση. Ε, συνιστόσα όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε και μια νέα εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να επεξεργαστούμε στα στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν πιστεύουμε ότι ε, αν υπάρχουν δεσμεύσεις σε εθνικό επίπεδο ε, θα έχουμε την κατάλληλη λύση. Πιστεύουμε ότι είναι πρόβλημα έλλειψης χρηματοδότησης. Ε, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν 25 δις ευρώ που προτείνονται για αυτή την πρωτοβουλία, πιστεύετε πραγματικά ότι θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Η πρόταση όπως έχει γίνει μας φαίνεται ότι είναι πολύ ρευστή, μια πρόταση η οποία είναι λίγο λογική για τα προβλήματα που έχουμε και θα θέσει και θέματα επικούρικότητα. Για να αποφύγουμε λοιπόν οποιαδήποτε παραβίαση τη αρχή τη Επικουρικότητα και της αναλογικότητας, οι εθνικέ, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει παρά το γεγονός ότι το επαναλαμβάνω συνεχώς, να είναι μόνιμος εταίρος για την ε, κατάρτιση και υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 21 Μαρτίου η Επιτροπή των ε, Περιφερειών θα εγκρίνει μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Είμαι συγχύτρια και η συγκεκριμένη διάσκεψη είναι μια πολύτιμη ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Εξονόμου. Αξαμίνου. Ε, Εξ Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής των Περιφερειών, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ που μας δώσετε το λόγο. Ε, θα τα ξαναπούμε του χρόνου, αλλά σας εύχομαι και μια καρποφόρα συζήτηση και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Uh, θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, ομιλητές για να απαντήσουν. Θα ε, ξεκινήσουμε με την αντίθετη σειρά, η Φαβιά Κέλ. Εγώ θέλω απλώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για τη συμμετοχή τους εδώ και να πω, Πρόεδρε, ότι αυτό που θα ήταν ωραίο θα ήταν στο τέλος των εργασιών μας να καταλήξουμε σε μια συνένεση που να εκφράζει μια κοινή πολιτική τοποθέτηση και ευχαριστώ την κυρία Μάρκες που αναφέρθηκε σε αυτή την ιδέα ψηφίσματος στο τέλος των εργασιών μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Για να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για να σταθμίσουμε τις διάφορες απόψεις. Και ξέρετε, η διάσκεψη αυτή δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει να πετύχει αυτή τη στάθμιση. Έχουμε πολλούς ομιλητές από τη δικιά μου πολιτική ομάδα, για παράδειγμα. Οπότε ευχαρίστω να αντικατοπτριστεί σε ένα κοινό κείμενο η δικιά μας η θέση, αλλά ή που θα πρέπει να ετοιμάσουμε κάτι πολύ γενικό με το οποίο συμφωνούμε όλοι και να μην χρειάζεται ψηφοφορία, αλλιώ αν χρειάζεται ψηφοφορία πώς θα σταθμίσουμε τις διάφορες απόψεις. Είναι πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μιλόσεβιτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Είναι προφανές. Το θέμα που μας απασχολεί όλους είναι οι κοινωνικές ανισότητες και η σύγκληση ε, στα κράτη-μέλη. Και συμφωνούμε όλοι. Μπορεί να μην ε, συμφωνούμε στους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές αυτές ανισότητες και πώς ακριβώς θα επιτύχουμε την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, συμφωνούμε, ε, συμφωνούμε όλοι ε, επί των στόχων και καθώς ε, προέρχομαι από τη δεξιά θα υπενθυμίσω τη βασική μου αρχή ότι πρώτα πρέπει να συλλέγει κανείς χρήματα και συνέχεια να τα δαπανά. Ο κ. Ζουγκέ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας τους ευρωβουλευτές να ακούμε τοποθετήσεις από τους εθνικούς βουλευτές το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι χρήσιμο. Μπορεί να φαίνεται ε, περίεργο να θέλουμε και να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Και εδώ θέλω να υπονομήσω αυτά που είπε η πρόσωπος Επιτροπής των Περιφερειών. Πράγματι, μόνο αν ενστενιστούν περισσότερο όλα αυτά οι εθνικοί βουλευτές, θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κρίστοφ Χάρτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι τοποθετήθηκαν για τα σχόλια. Και επειδή ε, υπερεξάντλησα το χρόνο μου στην αρχή δεν θα μιλήσω τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τάισεν, η Επίτροπος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε εξαίρετους διερμηνείς, οπότε, από ό,τι θυμάμαι τότε που ήμουνα και εγώ Ευρωβουλευτής, οπότε Ολλανδικά. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, αλλά πρέπει να απαντήσω σε κάποιε πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει που τέθηκαν προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, άκουσα πολύ καλά και σημείωσα τον όρο ενστερνισμός, ότι δηλαδή τον κύκλο αυτό του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να τον ενστερνιστούμε όσο γίνεται περισσότερο. Και έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, ε, με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης για την ανάπτυξη και για πρώτη φορά φέτος έχουμε αναλύσει πάρα πολύ με τις χώρες μέλη την έκθεση αναχώρα, περιμένοντας δηλαδή τις αντιδράσεις των χωρών μελών. Έχουμε συζητήσει με τις χώρες μέλη, με τις κυβερνήσεις. Ευχαρίστω να συζητήσουμε και με τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους. Είπαμε ότι οι επίτροποι κάνουν γύρω πάνε στις διάφορες πρωτεύουσε να συζητήσουν και ευχαρίστως να γίνουν συζητήσεις αυτές με τα εθνικά κοινοβούλια και βάσει όλων αυτών των συζητήσεων και βάσει των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των χωρών μελών και της δημοσιονομικής κατάστασης και θα καθοριστούν οι συστάσεις αναχώρα και θα συζητηθούν ε, με τους υπουργούς. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και φυσικά και θέλουμε να φροντίσουμε για τον ασθενισμό και τον ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια ώστε να γίνεται σωστά η ανάλυση και άρα και οι συστάσεις, οπότε να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, Χαίρομαι πολύ για όσα είπατε και την κοινωνική διάσταση που υπογραμμίστηκε ξανά και ξανά στη συζήτηση. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είμαστε πεπισμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται κοινωνική διάσταση στην οικονομία μας. Η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική πρόοδος πάνε χέρι-χέρι με την οικονομική πρόοδο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε μία οικονομία στην οποία να συμμετέχουν όλοι τότε θα είναι αποτελεσματική και ικανοποιητική. Και ο πυλώνας αυτός ο κοινωνικός πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπήρξαν και παρατηρήσεις για το ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Πράγματι. Και από την αρχή από τη θητείας της Επιτροπής αυτής με το σχέδιο Juncker όσον αφορά το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αυτό ακριβώ ήταν το σχέδιό μας, περισσότερες επενδύσεις και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να ενισχυθούν. Δεν είναι μόνο θέμα προπολογισμού, είναι θέμα και πού κατευθύνεται ο προπολογισμό μα. Από τη δικιά μα την πλευρά πάντω έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το περιθώριο ευελιξία. Ξέρετε ποιες είναι οι αποφάσεις που πήραμε ήδη τον Ιανουάριο του 2015. Ενισχύουμε λοιπόν την ευελιξία όσο γίνεται περισσότερο όταν χρειάζεται και τη ζουδούν οι χώρες μέλη. Και πρέπει να υπογραμμίσω και κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε, ότι η Eurostat είναι υπεύθυνη για την ταξινόμηση των διάφορων τμήματων του προπολογισμού. Είναι θέμα δικιάς μου αρμοδιότητας και πολύ χαίρομαι που η Eurostar έχει ετοιμάσει έναν οδηγό ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε τις επενδύσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα και μας λέει πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Έχουμε έναν οδηγό επίσης και για τις ενεργειακές συμβάσεις. Και είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε με τις κυβερνήσεις. Γιατί είναι κάτι που προσφέρει πολλές επενδυτικές δυνατότητες. Ρωτήσατε επίσης πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε όταν χρειαζόμαστε τόσες επενδύσεις στις οικονομίες μας, συγχρόνως να λέμε ότι χρειάζονται πολλές επενδύσεις και στον κοινωνικό τομέα. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Από τη δικιά μας την πλευρά πάντα μιλούσαμε για σύγχρονη κοινωνική προστασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν δίνουμε μόνο επιδόματα, αλλά η προστασία αυτή συνδυάζεται με υπηρεσίες που προσφέρει ο κόσμος και οι οποίες μας ενισχύουν ακόμα περισσότερο, μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα και έτσι οι άνθρωποι αυτοί εντάσσονται καλύτερα στην κοινωνία εφόσον έχουν αποκτήσει οι δυνατότητες και τους είναι πιο εύκολο στη συνέχεια να βρουν δουλειά. Αυτή είναι η επένδυση στον άνθρωπο που μας ανταμείβει στη συνέχεια και οικονομικά. Γι' αυτό μιλάμε για σύγχρονη μέθοδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ψηφιακή οικονομία σήμερα και ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Οι ανισότητες σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάθε χρόνο στις εκθέσεις χώρο, αναχώρα προσπαθούμε να δούμε πού βρίσκεται το θέμα των ανισοτήτων σε κάθε χώρα μέλος. Σίγουρα αυξήθηκαν οι ανισότητες με την κρίση, ακόμα Βέβαια όχι το ίδιο σε όλες τις χώρες, σε κάποιες χώρες έχουν μειωθεί οι κάτι που σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και να καταλήξουμε σε μια κοινωνία με τη συμμετοχή όλων. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για το ποια στοιχεία του κοινωνικού πυλώνα ε, θα ενισχύσουμε, ποιους νόμους προτείνουμε, τι προτάσεις γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποκτήσει σάρκα και οστά ο κοινωνικός πυλώνας, αλλά ίσως αυτά σε κάποια άλλη συζήτηση. Επίσης, ρωτήσατε για τα επίπεδα δανείων και τι γίνεται σε διάφορες χώρες όπου τα επίπεδα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Όντως, δύο συνεχόμενες χρονιές αναλύσαμε αυτό το θέμα και όταν ο δανεισμός είναι χαμηλότερος από την παραγωγικότητα, γίνεται η εξυπηρέτηση. Όταν όμως είναι το αντίθετο, τότε θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι συστάσεις πρέπει να κάνουμε και που τις κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια, ελπίζοντας να τις υλοποιήσουν οι χώρες μέλη. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πάντως και για τα προβλήματα με τις τράπεζες μετά την κρίση, αυτό εξακολουθεί να παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει βελτιωθεί κάπω η κατάσταση, η οικονομική ανάπτυξη βοήθησε σε αυτό, αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο πακέτο το οποίο αποτελεί βάρο στι οικονομίε μα. Τι πρέπει να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα πακέτο για να δώσει κάποιες προτάσεις στις χώρες μέλη όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αναγνωρίζουμε ότι οι συνέπειες για τους ανθρώπους είναι μεγάλες και ότι πρέπει να δείξουμε ευαισθησία στον άνθρωπο. Και δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι το έντις, που είναι η προστασία εγγύησης καταθέσεων. Προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο Συμβούλιο εξακολουθούν να υπάρχουν χώρες μέλη που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη βεβαιότητα, ε, να υπάρξει δηλαδή πρώτα μείωση του κινδύνου και μετά να υπάρξει ο επιμερισμός του κινδύνου. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε τώρα. Υπάρχει στο Συμβούλιο αυτός ο φάκελος για το έντι και συνεργαζόμαστε με τις χώρε μέλη για να δούμε πώς θα υπάρξει νέο δυναμισμός. Και τέλος, αλλά βέβαια αυτό μας φέρνει και σε άλλη συζήτηση, συνοχή. Ταμείο συνοχή πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι μια συζήτηση που εκρεμεί. Υπάρξει δημοσίες την προηγούμενη εβδομάδα της σχετικής έκθεσης και υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σενάρια τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στη διάσκεψη κορυφής. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να μειωθεί καθόλου ο προπολογισμό και ζητούν να υπάρξουν αρκετά μέσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί από το Brexit. Άρα πρέπει να βρεθούν χρήματα για να αντιμετωπιστούν κοινέ προκλήσεις, που είναι το προσφυγικό, μετανάστευση κτλ. Εδώ χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Με αυτό ολοκληρώνω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτήν και θα μεταφέρω τα όσα ακούσαμε εδώ σήμερα στους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή